Okay, dear colleagues, we should start. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Ας περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας, παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, εγκρίνεται. Σημείο δεύτερο στην ημερήσια διάταξη. Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην γραμματεία της Επιτροπής μας. Την 1η Οκτωβρίου, Εμιλιάνο Ημερώνη θα φύγει από τη γραμματεία της ΣΕΜΒΗ και θα αρχίσει να εργάζεται για τη γραμματεία της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω για την γενικότερη υποστήριξη που παρήχε στην εργασία των Ευρωβουλευτών και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα του θέση. Επίσης, να σας ενημερώσω για κάτι ακόμα όσον αφορά το καθεστώς διερμηνίας. Ο συνήθως έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες, χωρίς βέβαια εστονικά, λετονικά, μαλτέζικα και γκέιλικα. Όσον αφορά το web streaming και τα έγγραφα της συνεδρίασής μας, τα έγγραφα της συνεδρίασής μας είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-meeting και η συνεδρίασή μας θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου. Ας περάσουμε τώρα Στην πρώτη συζήτηση προβλέπεται στη μερίσια διάταξη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με το πρωτόκολλο για την εξάλληψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Αναμένω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το σημείο αυτό και ευθύ αμέσω θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Όστιν Ρόουαν είναι μαζί μας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 όπου εκπροσωπούνταν διάφορε γεωγραφικέ περιοχέ τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, προκειμένου να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο σε ε, προϊόντα καπνού. Στις, ε, το 2007 υποβλήθηκε η πρώτη αναφορά αυτής τη ομάδας εργασία και δημιουργήθηκε μία διακυβερνητική ομάδα διαπραγματεύση προκειμένου να συνταχθεί ένα κείμενο πρωτοκόλλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπηρεσίε των αρμοδίων γενικών διευθύνσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ συνεργάστηκαν έντονα για τα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν και υποβλήθηκε τελικά μια έκθεση για την COP5, την πέμπτη δηλαδή συνεδρίαση των μερών. Παρουσιάστηκε το κείμενο αυτό, εγκρίθηκε το κείμενο και ω τον Ιανουάριο του 2014 το κείμενο εκκρεμούσε ακόμα προκειμένου να υπογραφεί από τα κράτη-μέλη. Το 2013 υπογράψαμε εμεί το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο θα γίνει διεθνή συμφωνία μετά από την πάρα των 90 μερών αφορά τα μέρη υπογράψουν το πρωτόκολλο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ώστε το περισσότερο να υπογράψουν το πρωτόκολλο αυτό προκειμένου να γίνει ένα διεθνές νομικό όργανο για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνικών προϊόντων. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλουν έντονα στη διαδικασία αυτή. Έχουμε 29 μέλη, 28 κράτη-μέλη που συμμετέχουν και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ω ξεχωριστό μέλος. Σε λίγα λεπτά θα σας κάνω μια σφαιρική περιγραφή για το ποιο λόγο χρειαζόμαστε το πρωτόκολλο αυτό. Να δώσω όμως τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου Κορνίλιο Χόντμαρκ για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την επικύρωση από το Συμβούλιο του πρωτοκόλλου αυτού. Σε ευχαριστώ πολύ Όστιν. Το πρωτόκολλο αυτό για την εξάλληψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού είναι μια μεικτή συμφωνία, κοινή συμφωνία που σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να την υπογράψει αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία λοιπόν που σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει για το πώς θα μπορέσει εσωτερικά να υπογράψει το πρωτόκολλο αυτό, είναι η συμφωνία απόφασης, την οποία έχετε ενώπιόν σας. Σας υποβάλαμε το σχέδιο αυτό απόφασης, το υποβάλαμε και στο Συμβούλιο και συνεργαζόμαστε στενά με την Προεδρία του Λουξεμβούργου προκειμένου να εγκριθεί το κείμενο αυτό το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι στιγμή είχαμε τρει συνεδριάσει του Συμβουλίου αφιερωμένε στο ζήτημα αυτό και είμαστε πεπισμένοι ότι θα εγκριθεί πολύ σύντομη εν λόγω απόφαση. Σε ευχαριστώ, Κορνίλια. Τώρα, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε μια διεθνή συμφωνία για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση σε φόρους ή δασμούς που δεν καταβάλλονται και καταλαβαίνετε ότι αυτό επιβαρύνει τελικά και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους εθνικούς προπολογισμούς και το φαινόμενο αυτό το βλέπουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια άρα μιλάμε για 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε απώλειες όσον αφορά τον κοινοτικό και τους εθνικούς προπολογισμούς. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό είναι παγκόσμιο, χρειάζεται μια παγκόσμια λύση Οποιαδήποτε νομοθεσία και να χρησιμοποιήσει κανεί για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου εξαρτάται πάντα από την νομοθεσία που έχουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν καταρχάς για να ελέγξουμε την αλυσίδα εφοδιασμού. Στο τμήμα 3 του προτινούμενου πρωτοκόλου έχουμε συγκεκριμένα άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό, τη δέουσα επιμέλεια, τις ελεύθερες ζώνες συναλλαγών, τις πωλήσει αφορολόγητων ειδών, το ζήτημα του εντοπισμού και της παρακολούθησης. Ε, καταρχάς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό, για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση, άρθρο 8. Γιατί χρειαζόμαστε αυτό το άρθρο. Αν δούμε πώς είχαν τα πράγματα το 1998, βλέπουμε ότι ισχύουν ακόμα από τότε διάφορα πράγματα. Το 1998 είχαμε ένα σκάφος, το Envirana, το οποίο είχε πάνω του περίπου 55 με 6 φορτηγά, τα οποία μετέφεραν παράνομα τσιγάρα στην Ισπανία. Ξέρετε ότι σε κάθε από είχαμε 10.000 τσιγάρα. Χρειάστηκε λοιπόν να γίνει μια τεράστια διεθνής έρευνα με τη βοήθεια των ελληνικών και των ισπανικών λιμενικών αρχών. Καταφέραμε να εντοπίσουμε τον παραγωγό, ο βρισκόταν στην Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Βλέπαμε πάνω στο πακέτο ποιος ήταν βέβαια ο, κατασκευαστές, ο κατασκευαστής. Ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία Reynolds. Είδαμε ότι στη Βόρεια Καρολίνα βρισκόταν το εργοστάσιο αυτό. Είδαμε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο μηχάνημα το οποίο παρήγαγε αυτά τα τσιγάρα. Καταφέραμε να εντοπίσουμε ακόμα και τον χρόνο παραγωγής των τσιγάρων αυτών. Και τέλος καταφέραμε να βρούμε και το ίδιο το όνομα του μάνατζερ, του διαχειριστή ε, του εργοστασίου αυτού. Βέβαια η εταιρεία Reynolds μας είπε ότι δεν μπορούσε να δει τελικά σε ποιους πήγαιναν τα τσιγάρα αυτά, σε ποιους πολλούνταν παράνομα προφανώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στα πλαίσια της αλυσίδας αυτής εφοδιασμού να μπορεί κανείς να ελέγχει όλα τα στάδια από την παραγωγή, την κατασκευή των τσιγάρων μέχρι τον τελικό τους προορισμό. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε όλα αυτά τα άρθρα που έχουν να κάνουν με τον τοπισμό και την παρακολούθηση. Ένα άλλο άρθρο είναι η Δέουσα επιμέλεια. Πάλι η εταιρεία αυτή, η Reynolds, πολλούσε προϊόντα σε έναν μικρό πελάτη στην Γενέβη. 600 εκατομμύρια μάλλον πούλησαν τσιγάρα που αντιστοιχούσαν σε 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο και πάλι δεν μπορούσαν ακριβώς να εντοπίσουν ποιοι ήταν οι τελικοί τους ε, πελάτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να έχουμε ένα σύστημα εχνηλασιμότητας το οποίο είναι πιο, πολύ πιο αποτελεσματικό. Είναι πολύ σημαντικό όσοι πολλούν τσιγάρα να μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς σε ποιους πηγαίνουν αυτά τα τσιγάρα, ποιο είναι ο, ο τελικός προορισμός. Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η διεθνής συνεργασία πάλι είχαμε μια περίπτωση ότι παράνομη πώληση τσιγάρων μέσω της Ρήγα, τσιγάρα τα οποία πέρασαν στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τσιγάρα αυτά μέσω ουκρανικών φορτηγών θα κατέληγαν στην Αρμενία, αλλά τελικά σταμάτησε όλη αυτή η επιχείρηση στην Πολωνία. Καταφέραμε εκεί πέρα να δούμε ότι περίπου 70 κοντέινερ είχαν περάσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψιλοκομμένος καπνός, ο οποίο ουσιαστικά επιβάρεται από από τον ίδιο δασμό που παρήνει τελικά και τα τσιγάρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 77 εκατομμύρια ευρώ κανονικά έπρεπε να είχαν καταβληθεί στις τελωνιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάθαμε ότι ο καπνός αυτός προερχόταν τελικά από τη Βραζιλία, ήρθαμε σε επαφή με τους αρμοδίους στη χώρα αυτή, μπορέσαμε με τη δική τους τη βοήθεια να εντοπίσουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είχαν οργανώσει την παράνομη αυτή μετακίνηση καπνού, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάμε παραπέρα γιατί δεν είχαμε μία συμφωνία αμοιβαία συνεργασία και συνδρομής με τη Βραζιλία. Είδαμε ότι μόνο οι κάτω χώρες είχαν μια τέτοια συμφωνία δικαστική συνδρομής με τη Βραζιλία. Οι κάτω χώρες όμως δεν εμπλέκονταν στην όλη ιστορία, επομένω δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην έρευνα την οποία διεξάγαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, συντοπίσαμε τότε να έχουμε ένα σφαιρικό σύστημα διεθνούς συνεργασίας. Πιστεύω λοιπόν το πρωτόκολλο αυτό με όλες τις πτυχές του πραγματικά θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε και τη παράνομη αυτή πώληση τσιγάρων, αλλά καταφέρουμε να κτίσουμε επίσης και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία διαφεύγουν από τους εθνικούς προπολογισμούς. Σας ευχαριστώ και τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις από τους βουλευτές να σας πω ότι και η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΤΕ εκπροσωπείται στην αίθουσα. Επομένως, αν έχετε συγκεκριμένα ερωτήματα να απευθύνετε στους ανθρώπους της ΓΑΜΑ ΣΑΝΤΕ, ο κύριος ε, Ντομινίκ... Ε, η Ντομινίκ και ο Φιλίπ είναι εδώ για να σας απαντήσουν. Τρι, δύο βλέπω να έχουν στήσει το λόγο. Ο κύριος Καρχάνης Φλόρινς ο πρώτος. Äh, δεν έχω ξαναδεί επιτροπή με 11 εκπροσώπους τόσα χρόνια έχουμε εδώ. Καλός Ιωνός. Και μακάρι να εξελιχθεί και περαιτέρω. Από αυτό που είπατε για το πρωτόκολλο, για το λαθρεμπόριο, και το πότε κυρώθηκε. Φαίνεται να μην, ε, να μην μας είπατε ότι έχει κυρωθεί. Θέλετε να διευκρινίσετε λίγο περισσότερο. Για δε το είναι καπνοπαραγωγική αυτή η επιχείρηση. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Για να φανταστούμε ένας εισαγγελέα του Μιλάνου να προβαίνει σε συμφωνία με την ε, μαφία της Ιταλίας Δηλαδή διανοητικά δεν μου γίνεται αντιληπτό αυτό. Θέλετε να μου εξηγήσετε γιατί χρειάζεται μια συμφωνία. Εκτός και χωρίς να θέλω να είμαι επικριτικός, να μιλάμε για κάτι το πιθανό στο μέλλον. Μιλούμε για μια οδηγία, για τον καπνό. Είχαμε συνολικά καλά εργαλεία στα χέρια μας. Διεθνές πρωτόκολλο δεν έχει κυρωθεί. Γιατί λοιπόν πρέπει ειδικά με τη Φίλιπ Μόρις να προβείτε σε μια συμφωνία. Εμένα, για μένα είναι ένα βαρύτατο πλήγμα, κόλαφος αυτό το πράγμα. Τι έχετε να πείτε εσείς. Και έχουμε και τον εισηγητή εδώ της Επιτροπής μας. Αν θυμηθούμε το πώς η Φίλιπ Μόρις στράφηκε εναντίον μας και με πόσο αδυσόπιτο τρόπο μας έπληξε και τώρα πάμε να τους κάνουμε συμφωνίες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ίσως να έχω άδικο, ίσως να είναι διαφορετική η κατάσταση, ίσως εγώ να μην έχω καταλάβει. Και επίσης όλα αυτά τα χρήματα που πάνε. Όλα αυτά τα χρήματα που εισπράτετε, τι τα κάνετε. Και σε σχέση και με τα κράτη-μέλη, Φερρυπίν. στη Γερμανία, Φερρυπίν. Πού, σε ποιον πάνε τα λεφτά αυτά, τι χρηματοδοτείτε με τα χρήματα αυτά. Και περιμένω την απάντηση, εκτός και είναι τόσο περίπλοκο που θα χρειαστεί να μου τη δώσετε γραπτός. Ευχαριστώ, Πανιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάποιες διαπιστώσεις, πέντε τον αριθμό και τρεις ερωτήσεις. Γνωρίζουμε ότι το 12% των 6 δισεκατομμυρίων παράνομων τσιγάρων ε, μάλλον τσιγάρων ε, είναι ε, παράνομα και έχουμε και πάρα πολλά πραγματικά τσιγάρα 80% συγκεκριμένα άρα ποιος είναι αυτός ο οποίος ωφελείται δεύτερον ή τρίτον σίγουρα η καταπολέμηση του τσιγάρων είναι και το δημόσια υγεία πάνω απ' όλα. Όλοι συμφωνούμε, φαντάζομαι. Υπάρχει και διαφυγόν κέρδος, ε, το είπατε κι εσείς, εμείς ε, και το Κοινοβούλιο και εσείς το έχουμε υπολογίσει σε 12 δις ευρώ ετησίως. Άρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι το πιο αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης λαθρεμπορίου τσιγάρων είναι η χνηλασιμότητα η ανεξάρτητη όμως η χνηλασιμότητα ε, των παρέτων καπνού και γι' αυτό υιοθετήθηκε και το πρωτόκολλο το συγκεκριμένο. 54 κράτη στον κόσμο έχουν υπογράψει αυτό το πρωτόκολλο και στις 20 Δεκεμβρίου του 2014 το επέγραψε και η Ένωση. Και τρία κράτη μέλη μόνο το έχουν επικυρώσει αυτό το πρωτόκολλο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει το συντομότερο δυνατόν να έχουμε την επίσημη επικύρωση του πρωτοκόλου για την εξάλληψη του λαθρεμπορίου και για την ε, ε, δημιουργία πραγματικά ανεξάρτησης συνκλασιμότητας. Και έχω στα ερωτήματά μου η οδηγία για τα προϊόντα κάπνου που εγκρίθηκε το 2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 15 για την κλασιμότητα. Πώς συμβαδίζουν αυτά με το πρωτόκολλο της ΠΟΗ εάν και εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο ερώτημα. Το λαθρεμπόριο έχει αυξηθεί εντός Ένωσης κατά 30% τα έξι τελευταία χρόνια. Πώς εξηγείτε εσείς την αύξηση αυτή παρά το ότι έχουν συναυθεί συμφωνίες μεταξύ Ένωσης και ε, παρασκευαστών τσιγάρων ε, και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Και τρίτον, έχουμε διαπραγματεύσει για ενδεχόμενη επέκταση, το είπε και ο συνάδελφο Φλόρεντ, τη Συμφωνία Συνεργασία για την Καταπολέμηση τη Απάτη ε, με τη Philip Morris International 9 ναι, Ιουλίου του 2014 συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη εγκατέλειψαν την διαφορά νομική διαφορά ε, κατά της Philip Morris International με αντάλλαγμα συμφωνία η οποία συμπεριλάμβανε την καταβολή ενός 25 δις δολαρίων σε 12 χρόνια. Ε, θα λήξει σύντομα η συμφωνία αυτή. Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Θα προβούν σε μια αξιολόγηση και σε μια μελέτη αντικτύπου πρωτού προβούν σε κάποια μελλοντική ενδεχόμενη ανανέωση. Είμαι μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού και πρέπει να σας πω ότι ακούσαμε σε συνεδρία των θηρών την Επίτροπο το Φεβρουάριο και μας είπε η Επίτροπος ότι το Μάιο θα μας έδινε μία έκθεση αξιολόγησης. Ε, είμαστε Σεπτέμβριο και δεν έχω δει τίποτα ακόμη. Τώρα λοιπόν πλέον είναι κατεπήγον και δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας, είναι ε, ακόμη παραπάνω ε, αναγκαίο αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο, να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απαραίτητε ενέργειε. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημιουργήσουμε μια άτυπη ομάδα εργασία για την καταπολέμηση των παρεμβάσεων ε, της καπνοβιομηχανίας στα προϊόντα καπνού και θα είμαι πρόεδρος τη ομάδας. Ε, ευχαριστώ. Ε, κυρία Ριβασί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούστε, μας εξηγήσατε πόσο χρήσιμο είναι αυτό το πρωτόκολλο και εμείς είμαστε βέβαια υπέρ της κύρωσης του πρωτοκόλλου και από τα κρατημέλη και από την Ένωση. Λόγος είναι ότι θέλουμε να αυξηθεί διαφάνεια βέβαια. Και είπατε ότι έτσι θα ευνοηθεί και η διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητα Ταυτόχρονα όμως ε, τίθεται το εξή ερώτημα. Είπε και ο συνάδελφο Παγνιό, αυτές οι συμφωνίες, Αυτέ οι συμφωνίε με τη Φίλιπ Μόρι. τι θα γίνει με αυτές τις συμφωνίες. Είδαμε ότι επί σειρά ετών είχαμε αύξηση αυτού του λαθρεπορείου. Και βλέπετε πολύ καλό ότι να στήσουμε από βιομήχανο την κλασιμότητα ε, θα έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι από τη στιγμή που προέρχεται από το τσιγά, από, από μίμηση ε, έχουμε και κάποια χρήματα τα οποία ε, χάνονται από τα δημόσια ταμεία πώς θα τα δώσει αυτά στοιχεία ο βιομήχανος δίνεται το σύστημα, δηλαδή, μάλλον δίνει το σύστημα τη δύναμη στη φίλη που μόλι να πει όχι αυτά δεν είναι δικά μας τσιγάρα άρα δεν χρειάζεται να πληρώσουμε φόρους δεύτερον όταν ψηφίσαμε τον για τον καπνό Η Φίλιπ Μόρις ε, ετέθη αντίθετη προς αυτή την, ψήφα ψήφο των Ευρωβουλευτών. Από την ε, μία έχουμε τη Φίλιπ Μόρις, από την άλλη δεν έχουμε έναν ανεξάρτητο ε, φορέα για την χρηλασιμότητα. Ε, δεν πρέπει να ξεκάθαρα τα πράγματα. Και έχουμε και τις συμφωνίες αυτές. Ε, θέλω μια εξήγηση. Άλλο ερώτημα. Η όλα αυτή ρόλο παίζει εδώ μεταξύ μας. Η όλα αυτή έπρεπε να κάνει, έπρεπε να ελέγχει, να επαληθεύει αυτές οι επτά συμφωνίες με τη Φίλιππο Μόρις και τα κράτη και ερωτώ τι έκαναν για να δουν εκ του σύνεγγες και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αύξησης ε, του, της παραμυζιακίνησης. Ναι, είμαι υπέρ της κύρωσης πρωτοκόλλου και των ε, συμφωνιών αυτών, όμως γιατί αυτές οι συμφωνίες τελικά έχουμε κάποια σχέση με την καπνοβιομηχανία γιατί αυτό φαίνεται, δεν ξέρω. Κάποιο ταμείο ή κάτι άλλο θα πρέπει να σκεφτούμε. Και ήταν και στη συμφωνία, αλλά δεν το χρησιμοποίησαμε ποτέ. Αυτό το ανεξάρτητο Ινστιτούτο, ανεξάρτητο φορέα που θα έλεγχε τα τσιγάρα και δεν έγινε. Δεν συγκροτήθηκε αυτό ο φορέα, άρα υπάρχει και το ζήτημα του ελέγχου. Και θα ήθελα να τεθεί και το ζήτημα τη Όλαφ. Τσόφολη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το λαθρεμπόριο των τσιγάρων κοστίζει στους φορολογούμενους ε, πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μας το είπε αυτό ο μιλητής και κατά αυτόν τον τρόπο χάνουμε πάρα πολλά έσοδα, φορολογικά έσοδα. Ένα τσιγάρο στα 10 επίσης πέρυσι φάνηκε ότι προέρχεται από την παράνομη αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το συντομότερο δυνατό να καταφέρουμε να βρούμε λύσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο λύσεις που θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο και να φέρουμε, όπως είπα, σε ευρωπαϊκές και διεθνείς λύσεις, γιατί βλέπουμε ότι είναι διεθνείς οι δρόμοι που ακολουθεί το παράνομο εμπόριο και περνάνε ουσιαστικά από τη μία ήπειρο στην άλλη. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε μία λύση που θα διασφαλίζει καταρχάς την ασφάλεια των πολιτών, αυτών που καπνίζουν, και ας μην ξεχνάμε ότι το προϊόν αυτό είναι επικίνδυνο, δημιουργεί πάρα πολύ σημαντικές παθολογίες και τα νομικά μέσα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας τελικά δεν αποτελεσματικά, δεν τα κατάλληλα και δεν βοηθούν στο να καταπολεμήσουμε με τρόπο αποτελεσματικό το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ιδίως πέρα από τις δράσεις, τις ανακοινώσεις, τις δράσεις ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, θα πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως με τις νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν προκειμένου να βρούμε κάποιες καινοτόμες λύσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, όπως, όπως άλλωστε έχουν πει πάρα πολλοί που ε, δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να έχουμε ένα επίπεδο χνηλασιμότητας, το οποίο το έχουμε πετύχει για τα τρόφιμα. Τώρα θα πρέπει να καθιερώσουμε το ίδιο επίπεδο χνηλασιμότητας και για άλλα προϊόντα, όπως τα προϊόντα καπνού. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα και την προέλευση των προϊόντων αυτών η Ιταλία που είναι η πρώτη χώρα παραγωγή καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα τη χνηλασιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα θεμελιώδε προκειμένου να μην έχουμε ως το δυνατόν δυσμενεί συνέπειε για τους εργαζόμενους του τομέα αυτού που είναι περίπου 55.000 στην Ιταλία. Το δικό μου το ερώτημα έχει να κάνει κυρίως με το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει για την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου και αν τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα χνηλασιμότητας ή αν θα πρέπει τελικά να συνεχίσουμε να ζούμε με 28 διαφορετικά εθνικά συστήματα χνηλασιμότητας με όλους τους περιορισμούς και τα προβλήματα βέβαια που δημιουργεί με τέτοια κατάσταση. Ε, ε, ε, Βεβαίω, η προσπάθεια της ενίσχυσης της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καπνού είναι ευπρόσδεκτη, τη χαιρετίζουμε και ελπίζω να γίνει γρήγορα η διευκρίνηση και από τον Επίτροπο για διάφορα σημεία. Ε, με βάση το τίτλο 5 του τελευταίου τμήματος για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να μην είναι πλήρης θέση του Συμβουλίου. Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία καθώς και η ασφάλεια της Ένωσης απαιτούν να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία ορίζει και προτείνει το πρωτόκολλο. Επικαλούμε λοιπόν το άρθρο 67 παράγραφος 2 και την απουσία ελέγχου στα εσωτερικά της Ένωσης. Πώς θα ενισχυθεί ο αγώνας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού στην Ένωση αν η εσωτερική αγορά δεν ενισχυθεί με τα μέσα που έχουν θέση ε, μέσα στην επικράτεια του τα κράτη-μέλη. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, από τη διαπίστωση και των γαλλικών αλλά και των γερμανικών τελωνίων σημειώνεται σημαντική μείωση του προσωπικού στις δομές τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης και θέλω να υπογραμμίσω το ζήτημα της συνοχής ως προς τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εμπορικά ζητήματα, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, που υπογράφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, που συμφωνεί, που την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, σημαίνει πιο χαλαρή ε, παρακολούθηση των ε, ε, κινήσεων των εμπορευμάτων, κυρίως για τις χώρες διαμεσολάβησης. Η δε πώληση μέσω του ίντερνετ είναι ένα κύριο μέσον παράτυπου εμπορίου είναι δυνατόν να επιβάλλεται ή να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς της πωλής μέσω ίντερνετ με αυτό που ισχύει για την προσωπική αγοραπολισία, τη, με τη φυσική παρουσία. Επίσης, σε σχέση με την υιοθέτηση του πρωτοκόλου. τι είδους ερμηνεία μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τους όρους του που αναφέρονται στην επιμελητιακή αλυσίδα και τη δυνατότητα επέκτασης της στο εμπόριο δεδομένων των υποχρεώσεων για δέουσα επιμέλεια του άρθρου 7. Είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν αυτοί οι όροι στο ελληνικό εμπόριο. Το πρωτόκολλο. Βεβαίω καταλαβαίνω ότι έχει μια λογική για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού, αλλά δεν νομίζω ότι λύνει το προβλήματα. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί άλλο να λάβει το λόγο. Έχετε ερωτήσει. Εάν όχι, δίνω το λόγο στην Επιτροπή και πάλι. Ας ακούσουμε λοιπόν τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, άκουσα τις και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ας δούμε λοιπόν. Το φωνηθέν λοιπόν, κείμενο εγκρίθηκε το 2012 τον Νοέμβριο στη Σεούλ της Κορέας. Γιατί η κατάσταση των υπογραφών ήταν ανοιχτό έως τον Ιανουάριο του 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το υπέγραψε το Δεκέμβριο του 2013 και μέχρι τον Ιανουάριο που έκλεισε η προθεσμία για τις υπογραφές είχαν, κύρο, είχαν υπογράψει τέσσερα συμβαλόμενα μέρη εκ των οποίων ορισμένα έχουν ήδη κυρώσει, καθίσταται διεθνές νομοθέτημα 19 μέρες μετά την κύρωση από το 400 συμβαλόμενο μέρο. Σε αυτό το στόχο τίνουμε και πιέζουμε και αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να ασκήσουν το δυνατόν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σημαντικό επίσης και πρέπει να το αναφέρω ε, το σύστημα ανείχνευσης και παρακολούθησης της Φίλιπ Morris. Είναι το μόνο το οποίο έχουμε στη θέση μας αυτή τη στιγμή. Είναι το πρωτόκολλο προβλέπει η ανείχνευση και παρακολούθηση να ισχύει για πέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση της συνθήκης. Έτσι, ακόμα και αν έτοιμο στα τέλη του 2016, θα περάσουν πάλι πέντε χρόνια για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Επομένως, τι κάνουμε μέχρι τότε. η βασική ιδέα της ανείχνευσης και παρακολούθησης θα εντοπιστούν οι εγκληματίες. Το εξήγησα και νωρίτερα. Η συγκεκριμένη συμφωνία με τη Φίλιπ Μόρις και λοιπούς καποπαραγωγούς γιατί δεν πρόκειται για μνημόνια συνεννόησης αλλά για νομικά, δεσμευτικά και εκτελεστά κείμενα συμφωνίας που μπορούν να κρίνουν δικαστήρια. Έχουμε λοιπόν σημειώσει σημαντική πτώση στα νομότυπα προϊόντα τους από τη στιγμή που άρχισαν οι συμφωνίες, βέβαια δεν μπορούν να ελέγξουν το λαθρέο προϊόν και τίθε το ερώτημα, αφού το πρόβλημα εντείνεται, γιατί εντείνεται. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Αυτό οφείλεται στα λεγόμενα chip points, το γεγονό ότι παράγονται δηλαδή πάρα πολλά τσιγάρα σε διαφορέ τοποθεσίες ανά τον κόσμο και δεν μιλώ για το, λαφρέο, για το παραποιημένο προϊόν που έρχεται από την Κίνα κτλ. Αλλά για ζώνες ελεύθερων συναλλαγών με 17 συνολικά εργοστάσια και έλεγχο μηδενικό από τη στιγμή δηλαδή που παράγει το προϊόν δεν έχει κανένα πρόβλημα η σχετική διοικούσα αρχή. Αυτό το προϊόν έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο «Λοιπά προϊόντα». Μπορεί το πακέτο, να, ε, το κυβότιο να αναγράφει πάνω ε, μπλουζάκια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μέσα έχει τσιγάρα. Άρα, το πρόβλημα είναι βεβαίω το να λειτουργεί σωστά και λειτουργεί αυτή τη στιγμή η ανείχνευση και παρακολούθηση και όταν καταστεί ανεξάρτητο το σύστημα αυτό, και παρακολούθησης, όταν κυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη ε, το πρωτόκολλο, θα πρέπει να δεχθεί κάθε στοιχείο του πρωτοκόλλου και τις αναφορές στην ανέχνευση και παρακολούθηση, το γνωρίζουμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Για το TPD μπορεί ο συνάδελφος Σάντρα να βοηθήσει Παρακαλώ, αυτό το λόγο. Ευχαριστώ, στην. Χαίρομαι πάρα πολύ που επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Έμβη, όπου κατά το παρελθόν συζητήσαμε και διαπραγματευθήκαμε διαμακρών ε, την οδηγία για το πρώτο καπνού. Χαίρομαι πραγματικά. Δύο ερωτήσεις νομίζω απευθύνονταν ε, στην τίζη, στην ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΤΕ. Το ένα αφορούσε τη σχέση μεταξύ του άρθρου 15 και του πρωτοκόλλου περί λαθρεμπορίου. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι κατά την άποψή μας το άρθρο 15 και το πρωτόκολλο περί λαθρεμπορίου είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Το άρθρο 15 θεσπίζει ένα σύστημα ανείχνευσης ε, και ιχνηλασιμότητας για τα πρώτα παράγονται στην Ένωση και προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Το ίδιο κάνει και το πρωτόκολλο περί λαθρεμπορίου που βέβαια πάει λίγο πιο πέρα σε κάποιες πτυχές. Όμως, ε, όπως είναι η διεθνής ε, προστασία που δεν προβλέπεται στο άρθρο 15. Όμως αυτό κατά την άποψή μου είναι και αυτονόητο. Τώρα, θεωρούμε ότι από τη στιγμή που το άρθρο 15 μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και υλοποιηθεί από τα κράτη-μέλη, θα έχουμε πλέον συμμορφωθεί προς ε, την υποχρέωσή μας ε, για υποχρέωση του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου περί λαθρεμπορίου, κάτι που είναι ένα πολύ θετικό, πολύ καλό βήμα για τη διεθνή κοινότητα. Τώρα, δεύτερο σχόλιο. Σχέση του άρθρου 15 πάντα και πρωτοκόλλου περί Πού βρίσκεται η εφαρμογή του άρθρου 15 μέχρι τώρα. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν το σύστημα εντοπισμού και χνηλασιμότητας, ανείχνευσης, ε, μέχρι το 2019, Μάιο του 2019 είναι επιχειρησιακό. Τι κάναμε λοιπόν, ε, από το 2013 ήδη ξεκινήσαμε τη μελέτη σκοπιμότητας που δείχνει ότι είναι δυνατόν να έχουμε εντοπισμό και ανείχνευση εντός Ένωσης. Βέβαια είναι λίγο πιο πολύπλοκο αυτό σε σχέση με το τι θα κάνουν τα συμβαλόμενα μέρη στο πρωτόκολλο, γιατί υπάρχει διασυνοριακό εμπόριο εντό Ένωση, άρα πρέπει να δούμε το διασυνοριακό εμπόριο, να αντιμετωπίσουμε τα σχετικά ζητήματα. Έχουμε επίση ε, προχωρήσει και σε μια πρώτη σειρά διαβουλεύσεων για τη μελέτη τη σκοπιμότητα και θα ξεκινήσει, ξεκινά ήδη η δεύτερη μελέτη τη σκοπιμότητα. Προβλέπεται στο άρθρο 15 και εφαρμοστική νομοθεσία των ε, το καλοκαίρι του 2017 θα είναι έτοιμη και θα, δεις, θα δώσει δύο χρόνια προθεσμία στα κράτη-μέλη και στην βιομηχανία περίπου για να υλοποιήσουν το σύστημα ελέγχου ε, ανείχνευσης μάλλον και ε, αυτό θα πρέπει να είναι όπως είπαμε το 19 ε, να ισχύει αυτό το σύστημα για τον καπνό και πέντε χρόνια μετά για τα υπόλοιπα προϊόντα καπνού. Αυτά για τη σχέση μεταξύ πρωτοκόλλου και άρθρο 15. Και επειδή έχω και το μικρόφωνο, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω ένα ακόμη σχόλιο τέθηκε ένα ερώτημα τι κάνουμε με το διαδικτυακό εμπόριο, τις διαδικτυακές πωλήσει, ε, που είναι μια σημαντική πτυχή, ή ήταν αυτή η ερώτηση, είναι μια σημαντική πτυχή ε, στο το μέτωπο του λαθρεμπόριου. Πράγματι είναι, είναι η απάντηση. Το διαδικτυακό εμπόριο, οι διαδικτυακέ συναλλαγέ βέβαια αντιστοιχούν σε ένα πολύ μικρό κομμάτι των πωλήσεων εντό Ένωση και αυτό διότι πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν λάβει μέτρα κατά των διαδικτυακών πωλήσεων. Δύο σχόλια. Πρώτον, πάλι ότι σίγουρα θα καλύπτονται οι διαδικτυακές πωλήσει ε, από τα μέτρα ε, εντοπισμού και ανείχνευση δεν απολύεται κανένα προϊόν δηλαδή στην Ένωση αν δεν ισχύουν αυτά τα μέτρα, το ίδιο ισχύει για το διαδίκτυο. Δεύτερον, τα προϊόντα καπνού, η οδηγία για τα προϊόντα καπνού προβλέπει τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη είτε να απαγορεύσουν ε, τις διαδικτυακές ε, πωλήσει συνοριακά ή γενικώ, είτε να υιοθετήσουν ένα αυστηρό καθεστώς ελέγχων όπου ο προμηθευτής πρέπει να έχει ε, την έδρα του ε, στη χώρα προέλευσης και θα πρέπει και στη χώρα ε, προορισμού να μπορεί να παληθευτεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες για την παραγωγή αυτών των τσιγάρων. Ο κύριος Γκρέτη θέλει το λόγο. Ναι. Είναι καλό ότι υπάρχει αυτή η υλοποίηση, η αξιολόγηση υλοποίηση εδώ στο κοινοβούλιο γιατί αφιερώνουμε κάποιο χρόνο από το πρόγραμμα της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό. Γιατί νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και στο επόμενο θέμα, πώς υλοποιείται δηλαδή η οδηγία πλαίσιο. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται και αντιμετωπίζεται βέβαια η νομοθεσία του συνάδελφος Φλόρεντς <laughs> το ανέφερε με την ε, μεγάλη εκείνη εκδήλωση για την οδηγία για τα προϊόντα καπνού που ήμουν υπεύθυνο και εγώ ως πρόεδρος αλλά και στα θέματα που είχαν να κάνουν με τις εκπομπές οξύδου του άνθρακα και τους κύκλους δοκιμών ήταν πολύ σκληρές ε, διαπραγματεύσεις και συστήσεις αλλά δεν είδαμε τίποτα σαν αυτό που ήταν στην υπόθεση του καπνού από τις μεγάλες επιχειρήσεις που αναφέρατε κι εσείς. Είναι λοιπόν αδιαφανή τα λόμπι αυτά, πολύ αδιαφανή και κυρίως θέλω να αναφερθώ στη διάθεση μέσω του ίντερνετ και επίσης στη διάθεση ενός άλλου τύπου προϊόντος που είναι τα υγρά για τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα. Τι γίνεται στην υπόθεση αυτή, υπάρχει κάποια ρύθμιση. υφίσταται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή εναπόκειται στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία. Ήταν ένα πολύ διαφιλονικούμενο ζήτημα όταν συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο μέλλον τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα. Και σε ποια κατηγορία θα πρέπει να υπαρθεί το σχετικό εμπόριο, γιατί Ξέρουμε ότι πολλά από τα σχετικά υγρά προέρχονται από την Κίνα. Ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι η Κίνα έχει τις ίδιες, το ίδιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας ε, για τα, σχετικά, για τα υγρά των ηλεκτρονικών σιγάρετων όσο έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Περιμένω λοιπόν να ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας και νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο και να κάνουμε συζητήσεις πολύ πιο τακτικά. Δεν, είναι, δεν πρέπει να είναι δηλαδή μια συμπτωματική ε, συζήτηση αυτή που αφορά τον τρόπο εφαρμογή τη νομοθεσία είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθεί τακτικά το Κοινοβούλιο. Η εφαρμογή, η υλοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση τη κάθε νομοθεσία, στην κάθε περιοχή πρέπει να εξετάζεται από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και η κυρία Ριβαζή που θα ήθελε να δει το λόγο. και μετά θα μιλήσει η Επιτροπή. Η κυρία Ριβάζη λοιπόν σύντομο σχόλιο και επιστρέφουμε στην Επιτροπή. Για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχα μια ερώτηση για το ρόλο της ΟΛΑΦ και εκεί απάντηση δεν μου δώσατε. Στο πλαίσιο των συμφωνιών με τη Φίλιπ Μόρις, 80% από τα έσοδα πάνε στα κράτη-μέλη, 9,7% δε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πού πάνε τα λεφτά αυτά, πώς αξιοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, που διαπιστώνεται ότι ενισχύεται, ενώ έχετε διανύμητα τόσο χρήμα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Θέλουμε τη διαφάνεια από αυτό. Ευχαριστώ και τώρα η Επιτροπή και πάλι. Έχετε λόγο. Oh, no, um, okay, Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού απαντήσω το ερώτημά σα αυτό σε σχέση με τις πωλήσει στο διαδίκτυο. Να συμπληρώσω και εγώ αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Ντομινίκ. Οι διαδικτυακές πωλήσει θα υπαχθούν και αυτές σε όλες εκείνες τις διατάξεις που έχουμε στο πρωτόκολλο και επομένω θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανεί τέτοιε πωλήσει. Θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώ ποιο είναι ο πελάτη και θα πρέπει ο κατασκευαστή να είναι σε θέση να εντοπίζει και να παρακολουθεί του πελάτε αυτού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για τι πωλήσει αυτέ τα ίδια μέσα που έχουμε για τι συμβατικέ πωλήσει. Όσον αφορά την Όλαφ, ο συνάδελφός μου, Γεώργ Ρέμπλινγκ, θα σας πει περισσότερα πράγματα όσον αφορά αυτό το 90% που πάει στα κράτη-μέλη και το 9% των εσόδων που πάει στα κράτη-μέλη. Τα χρήματα που πάνε καταρχάς στο κοινοτικό προπολογισμό πάνε άμεσα στον κοινοτικό προπολογισμό. Δεν είμαι η Δήμων, δεν προέρχομαι από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού, αλλά πάρα πολλές φορές μας έχουν πει ότι δεν γίνεται να πούμε ακριβώς πού θα πάνε τα χρήματα αυτά, να δεσμευθούν για συγκεκριμένε δράσει. Σε ορισμένε περιπτώσει κάποια κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, αλλά βέβαια τα χρήματα αυτά σε κάθε περίπτωση καταλήγουν στα Υπουργεία Οικονομικών, τα οποία αποφασίζουν πώ θα διαθέσουν αυτά τα χρήματα. Πάντω καταλήγουν με τον έναν άλλο τρόπο τα χρήματα αυτά στου εθνικού προπολογισμού. Για παράδειγμα, η Αυστρία έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά προκειμένου να χρηματοδοτήσει όλες αυτές τις δράσεις κατάσχεσης παράνομων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα κράτη-μέλη αποφασίζουν αυτά πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα αυτόνομα, ανεξάρτητα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε να συμπληρώσω τα όσα είπε ο και σε σχέση με τις ερωτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοί σας. Είμαι αρμόδιος της Όλαφ ε, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, ονομάζομαι Γκέωρκ Ρέμπλινγκ δεν μπορούμε, όπως καταλάβατε, με ένα μόνο μέτρο να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Χρειάζονται πάρα πολλές πρωτοβουλίες προκειμένου να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό στο σύνολό του. Από τις 30 Ιουνίου όμως του 2015 έχουμε πλέον μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Εφαρμόζουμε τη στρατηγική αυτή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα των πιο βασικών σημείων αυτής της ανακοίνωσης και της στρατηγικής. Βασική μας προτεραιότητα είναι καταρχάς η κύρωση του πρωτοκόλου. Το συζητήσατε αυτό πριν από λίγο. Αυτό αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και για μας προκειμένου να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο πρώτων καπνού. Συνεργαζόμαστε βέβαια με τους αδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όλε οι διατάξει εντοπισμού και παρακολούθηση όπω προβλέπονται στην οδηγία προϊόντων καπνού. Παράλληλα όμω, γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με το ζήτημα τη εφαρμογή νομοθεσία, Ο αριθμό των κατασχέσεων από τα κράτη-μέλη έχει μειωθεί και μειώθηκαν σημαντικά ιδίω όσον αφορά τι ε, κοινοποιημένε κατασχέσεις ε, από εταιρείε τα τελευταία χρόνια τα κράτη-μέλη, οι αρχές κατάσχεσης μάλλον των κρατών μελών έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 από την Φίλιπ Morris 60 εκατομμύρια τσιγάρα, αριθμός ο οποίος μειώθηκε στα 30 εκατομμύρια. Επομένως, ο αριθμός του κατεσχόμενου καπνού ουσιαστικά έχει μειωθεί σημαντικά. Δημιουργήσαμε πάντως και ένα νέο εργαστήριο προκειμένου να μπορούμε ανεξάρτητα να αναλύουμε τα τσιγάρα τα οποία έρχονται στην δική μας την την ιδιοκτησία. Συνεργαζόμαστε πάλι με τα κράτη-μέλη. Ολοκληρώσαμε πρόσφατα μία επιτυχή συνεργασία με τα κράτη-μέλη στην περιοχή της Βαλτικής. 13 εκατομμύρια τσιγάρα καταφέραμε να κατασχέσουμε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτό το μήνα μία πρωτοβουλία της όλα που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είδαμε ότι δόθηκε η έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλετε κι εσείς όπως είδα να τροποποιηθεί η ε, οδηγία 515 κάτω 97 για την καταπολέμηση της ε, φορολογικής ε, τελωνιακής απάτης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που εγκρίθηκε η σχετική πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αυτό μας δίνει τελικά νέα μέσα, νέα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού. Όσον αφορά τη Φίλιπ Μόρις, ακούσαμε πολλά ερωτήματα για το τι θα γίνει στο μέλλον. Όπως είπατε πολύ σωστά, θα, θα τελειώσει η ισχύ της συμφωνίας αυτής τον Ιούλιο. Καλούμεθα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Είμαστε σε επαφέ με τα κράτη-μέλη, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η δική τους εμπειρία από την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Θέλουμε να δούμε και ποια είναι η εμπειρία από την εθνική εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια αξιολόγηση της εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, η οποία θα κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατό αφού του οριστικοποιηθεί. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αν θα ζητήσει παράταση της συμφωνίας αυτής. Αυτή τη στιγμή προφανώς δεν γίνονται διαπραγματεύσεις και ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να εξετάσουμε είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, το ότι η κατάσταση σήμερα διαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με αυτή που είχαμε πριν από 15-20 χρόνια. Έχουμε πλέον την οδηγία για τα πρώτα καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον θα έχουμε σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το διεθνέ αυτό όργανο, το πρωτόκολλο. Πρέπει όλα αυτά να λεφθούν υπόψη στην αξιολόγηση τη συμφωνία με την Φίλη Πόρη, η οποία θα διεξαχθεί πολύ σύντομα και προφανώ το πόρισμα τη αξιολόγηση αυτή θα στο κοινοποιήσουμε το στομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν η Γενική Διεύθυνση Σάντετ θέλει να πάρει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για το άρθρο 20 έθεσα ένα ερώτημα για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Να απαντήσω. Όπως γνωρίζετε όλοι το άρθρο 20 φέρει, αν θέλετε, ε, την υπογραφή του Κοινοβουλίου, γιατί αυτό είχε την ιδέα να αντιμετωπιστούν αυτά τα προϊόντα ως καταναλωτικά αγαθά. Μας πείσατε τότε ότι θα πρέπει να διαπόμεθα από τρεις αρχές. Η πρώτη είναι ότι τα προϊόντα που διατίθεται στο εμπόριο πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας. Δεύτερη αρχή να μην είναι ελκυστικά για την νεολαία, αλλά για τους καπνιστές που θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα και όχι για ανθρώπους ε, που ξεκινάνε ε, να καπνίζουν με ηλεκτρονικά τσιγάρα και εθίζονται στην νοικοτήνη και τελικά καταλήγουν να γίνουν καπνιστές μεταγενέστερα. Και τρίτη αρχή, ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα νέα προϊόντα, διότι έρχονται σε τακτά διαστήματα στη δημοσιότητα νέε επιστημονικές μελέτες, αλλά και νέα προϊόντα βγαίνουν στην αγορά τακτικά ε, και πρέπει να τα παρακολουθούμε. Να παρακολουθούμε όλε αυτέ τι εξελίξεις. Χαίρομαι ε, πολύ που μπορώ να πω ότι όλα τα κράτη-μέλη με τα οποία έχουμε πολύ καλές ε, επαφές εργάζονται σκληρά για την μεταφορά τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο και προσπαθούν επίσης ε, να εφαρμόσουν πιστά και το άρθρο 20. Για παράδειγμα υπάρχουν κανόνες ε, για τις ε, διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσει για τα προϊόντα καπνού και υπάρχει, όπως και για τα προϊόντα καπνού μάλλον, και γίνονται διάφορες σκέψεις το αν πρέπει να επιτρέπονται να απαγορευθούν. Επίσης υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όπως ξέρετε, για το τι μπορεί να κάνει ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, τις πωλήσεις προς ανήλικους. Αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα και τώρα πολλά κράτη-μέλη πάνε πιο μακριά και ε, εξετάζουν το ενδεχόμενο πώς να ρυθμίσουν ε, αυτό το θέμα ή ε, για το πώς θα μπορεί να υπάρχουν ε, χώροι ε, απαλλαγμένοι από καπνό ή τα τσιγάρα που δεν ρυθμίζονται από την οδηγία, τα οποία δεν περιέχουν νοικοτήν, για παράδειγμα. Επίσης και η Κομισιόν εργάζεται για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, για τα επαναπληρώσιμα συγκεκριμένα, τις επαναπληρώσιμες συσκευασίε. Θέλουμε να δούμε επίσης τι κίνδυνοι προκύπτουν με την διαδικασία αυτή της ε, όταν δηλαδή έχουμε ανταλλακτικά και τα ξαναγεμίζουμε και θέλουμε περισσότερα στοιχεία από τους εισαγωγείς και τους ε, παρασκευαστές ηλεκτρονικών τσιγάρων. Είμαστε σε καλό δρόμο με την υλοποίηση θα έλεγα. Αν έχετε περισσότερα ερωτήματα μπορούμε να επανέλθουμε κάποια στιγμή εδώ. Δείτε και την ιστοσελίδα μας, έχουμε ένα σχέδιο υλοποίηση για όλα τα μέτρα που θα λάβουμε πριν το Μάιο του 2016 και προς το παρόν τηρούμε πιστά το χρονοδιάγραμμα, όπως για παράδειγμα οι εκτελεστικές πράξεις για την επισήμανση θα εγκριθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και έτσι η βιομηχανία θα έχει πολύ χρόνο μπροστά τη ε, μέχρι το Μάιο του 2016 για να προσαρμόσει τις διαδικασίες παραγωγής της, ε, στις νέες ε, ε, στους νέους κανονισμούς συσκευασίας. Ε, τις επόμενες δύο εβδομάδες ε, θα τα έχουμε αυτά, άρα έχουν 6-7 μήνες μέχρι το Μάιο του 2016 στις βιομηχανίες. Αυτά ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Καιρό, όχι, είμαι εντάξει. Ο πρόεδρος, να σας ευχαριστήσω τότε όλους και του εκπροσώπου τη Όλαφ και του εκπροσώπου τη ε, ΓΑΜΑ ΣΑΝΤΕ που ήρθατε εδώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων ε, και την ε, αυτή η ενημέρωση για το πρωτόκολλο καταπολέμηση του λαθρεμπορίου του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση, ήταν, δεν ήταν όμω και τελευταία. Η συζήτηση θα συνεχιστεί όχι μόνο στην Επιτροπή μα αλλά και σε άλλες επιτροπές. Όσο συνεχίζουμε το έργο μας σε αυτό το σημαντικό τομέα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που συμμετείχατε στη συζήτηση και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης και δίνω ξανά τη σκητάλη στον πρόεδρό μας τον κύριο Λαβία. Okay, we can uh, continue the next Συνεχίσουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, παρουσίαση της έκθεσης EPRS με θέμα έκθεση σχετικά με το κόστος της μη ολοκλήρωσης Ευρώπης όσον αφορά την νομοθεσία για τα ύδατα. Έχουμε εδώ τη Γενική Διεύθυνση Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δίνω το λόγο στον κύριο Τζο Ντάν, ο οποίος είναι υπηρεσιακός διευθυντής της EPRS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ντάν ονομάζομαι και είμαι υπηρεσιακός διευθυντής ε, για τις μελέτες αντικτύπου και την προστιθέμενη αξία στη Γενική Διεύθυνση EPRS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πρώτη φορά που παίρνω το λόγο στην Επιτροπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεται να κάνω μια παρουσίαση και εδώ, καθότι έχω πάει και σε άλλε επιτροπέ του Κοινοβουλίου, δεν είχα έρθει ακόμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Βασική μα αποστολή είναι να καταφέρουμε να δίνουμε σε επιτροπέ τα απαραίτητα μέσα παρακολούθηση και εντελεχού έρευνα, ιδίω όσον αφορά κυρίω τι μελέτε αντικτύπου που γίνεται εκ των προτέρων και των εκ των υστέρων σε σχέση με την εφαρμογή κοινοτική νομοθεσία. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα μέσα ποσοτικοποίησης και χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα μέτρα μέτρησης της απουσίας της Ευρώπης τελικά, της απουσίας κοινοτική νομοθεσίας σε σχέση με διάφορους τομείς και θέλουμε να μπορούμε χρηματικά, οικονομικά να ποσοτοκοποιούμε κάπως επιπτώσεις αυτές. 1,6 εκατομμύρια ευρώ περίπου θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν αν είχαμε περισσότερη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όσο περισσότερο ερευνούμε τα ζητήματα αυτά, τόσα περισσότερα κέρδη διαφεύγοντα ουσιαστικά καταφέρνουμε να εντοπίσουμε. Σήμερα παρουσιάζουμε μία μελέτη την οποία μας ζήτησε η προηγούμενη θητεία της δικής σας επιτροπής όσον αφορά την ομοθεσία για τα ύδατα. Θέλαμε πάλι να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής ο κύριος Ζέιμπορ ήταν τότε εισηγητής για το ζήτημα αυτό και στην συνάντηση που είχα με τους συντονιστές σας στην προηγούμενη νομοθετική θητεία μου είχε συζητηθεί να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα ζητήματα της εφαρμογή, ζητήματα της εφαρμογής της νομοθεσίας όσον αφορά τα ύδατα. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν η αξιολόγηση αντικτύπου, να κάνουμε μία ανάλυση κόστους-οφέλους και γι' αυτό το λόγο λάβουμε υπόψη Μα το κόστο τη εφαρμογή υλοποίηση, ε, το διοικητικό άκθο το οποίο προκαλεί ενδεχομένω η εφαρμογή τη κοινωτικής νομοθεσία. και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε μέσω τη κοινωτικής δράση 2,8 δισεκατομμύρια ετησίω. Πριν το καλοκαίρι θα διαβιβάσαμε κάποιες γραφικές ε, παραστάσεις και ή δυνατόν θα ήθελα τώρα να δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες οι οποίοι συνέταξαν την έκθεση αυτή. Θα ήταν καλό να σας παρουσιάσουν το πόρισμα της έκθεσης αυτής, αλλά δυνατόν να δούμε επίσης και ένα σύντομο βίντεο 4 λεπτών που συνοψίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα στο παρελθόν, ελπίζω να καταφέρουμε να δούμε τώρα τους αγγλικούς υπότιτλους και θα συμπεριλάβουμε και άλλες γλώσσες στη συνέχεια, όπως τα γαλλικά και τα γερμανικά. Ας δούμε δυνατόν λοιπόν κύριε Πρόεδρε το σύντομο αυτό βίντεο και στη συνέχεια δυνατόν να δώσουμε το λόγο και στους εμπειρογνώμονες που συνέταξαν την έκθεση. Και προφανώς είμαστε στη διάθεσή σα και για να απαντήσω ερωτήσεις, Πρόεδρος. Ας δούμε όντως το φιλμάκι αυτό και στη συνέχεια θα ακούσουμε και του συντάκτε τη έκθεση.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 This way, the EU would save billions of cubic meters of water and save approximately 25.8 billion euros annually. Thank you for... Σας ευχαριστώ για την ταινία. Και τώρα... Ο κύριος Στέφαν Σόιερ και ο κύριος Βίλιαμς για την παρουσίασή τους. Ευχαριστώ πολύ. Rob Williams. Μια σύντομη παρουσίαση. Στα θέματα που αρχίσατε να διαρευνήσουμε, εξηγούμε τη μεθοδολογία μας, εκθέτουμε τα ζητήματα. Αναπτύσσουμε λίγο αυτά που είδατε και στην ταινία και ο Στέφαν μετά θα σας παρουσιάσει τα ευρήματά μας τα πιο ενδιαφέροντα. τι κληθήκαμε να κάνουμε, όπως είπε και ο Τζον. Μία εξπόστη και μία εξάντε αξιολόγηση, μελέτη. Κοιτώντα ε, προς τα πίσω, μελετήσαμε την υλοποίηση της φυστάμενης νομοθεσίας για τα έδατα. Κοιτώντας προς τα μπρο προς το μέλλον, εκτιμούμε το κόστος και τα ωφέλη από την κάλυψη όποιων κενών μπορεί να υπάρχουν στην υλοποίηση. Και βέβαια περισσότερο κοιτάξαμε το τι ισχύει μέχρι τώρα, προς τα πίσω δηλαδή ιστορικά, καθώς είναι πιο πολλά τα διαθέσιμα δεδομένα και το υλικό που είχαμε να επεξεργαστούμε. Σύντομα θα σας εξηγήσω τη μεθοδολογία μας. Μελετήσαμε την φιλολογία που υπάρχει, αρκετό υλικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιολογήσεις συνεπειών, περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, αξιολογήσεις φυσταμής νομοθεσίας, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Πολλές μελέτες δείχνουν πώς ε, εφαρμόζουν ε, και τι συμπληρωματικό έχουν κάνει. Πήραμε υλικό από μη κυβερνητικέ οργανώσει, από πανεπιστήμια, ώστε να δούμε περισσότερο υλικό μπορούσαμε να μελετήσουμε. υλοποίηση μέχρι σήμερα. Αρχίσαμε να περιγράφουμε το περιβάλλον, το εδάτινο περιβάλλον και τους αφούς κύκλους του νερού, ώστε να δούμε αν η κάλυψη είναι επαρκής, η κάλυψη της ομοθεσίας, δηλαδή καλύπτει όλο τον κύκλο και αν υπάρχει κάποιο σημαντικό κενό που χρειάζεται προσοχή. Επίσης, κοιτάξαμε τις διάφορες οδηγίες τι προέβλεπαν, τι είχε πραγματικά συμβεί, τι είχε γίνει. Και αυτό με βάση και τις εκτιμήσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και άλλων φορέων. Σημαντικό κομμάτι στην προσέγγιση μας ήταν η σύγκριση της δικής μας προσέγγισης με το λεγόμενο blueprint της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. του προσχεδίου δηλαδή αξιολόγησης όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε σημειώσει πως για το 2020 θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια επαναξιολόγηση και να αφιγραμμιστούν οι προσπάθειες σχετικές με τους ε, επιδιωκόμενους στόχους για τα ύδατα, γιατί όπως λέει και η ταινία μας δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη πρόοδος. Κοιτώντας προς το μέλλον, προς τα μπρος, σε τρεις συγκεκριμένους τομείς με πέντε πρακτικά θέματα όπου προσπαθούμε να περιγράψουμε σημεία στα οποία θεωρούμε πως υπάρχουν προβλήματα, κενά στην υλοποίηση και πιθανά προβλήματα. Πολύ απλά θα ήθελα να εξηγήσω τα κύρια ζητήματα. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα εισήφθη το 2000 και άλλαξε την πραγματική φύση της οδηγίας για τα είδωτα, το πεδίο εφαρμογή, την κάλυψη και ξεπέρασε την ε, παρουσία του ανθρώπου στον ανθρώπου στον κύκλο του νερού αλλά και ολόκληρο τον ε, κύκλο του νερού με προσέγγιση ως προς τις ε, κοίτες των ποταμών που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και που πρέπει να εξετάζονται ως σύνολα και όχι ως τμήματα που ανήκουν σε διαφορετικές επικράτειες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο ήταν η προσέγγιση σε σχέση με την κατάσταση των υδάτων, την καταγραφή, την απογραφή της κατάστασης το 2015. Συγκεκριμένα τρία κύρια σημεία εκτίμησης, η ποιότητα, παρουσία δηλαδή ρήπων, ζυζανιοκτώνων, χημικών, αλλαγή θερμοκρασίας λόγω φερρυπίν ε, υδάτων που χρησιμοποιούνται στην ψήξη των πυρηνικών εργοστασίων, ε, ελάχιστες ανώτατες ροές, διαθεσιμότητα του ύδατος ως πόσιμου ή για άλλες χρήσεις και τρίτο τμήμα η χωρική προσέγγιση, δηλαδή οι εξελίξεις ως προς την παρουσία των ε, και η γεωφυσική ε, στις κοίτες των ποταμών και τη συνέχεια τους. Εδώ θέλω να σας δείξω την κάλυψη από διάφορες οδηγίες που εξετάσαμε κάτω δεξιά βλέπετε το διαχωρισμό μεταξύ χώρου και ποιότητας και ποσότητας, δηλαδή το καθεστώς, όπου στην ποιότητα έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο οδηγιών. Η οδηγία πλαίσιο για τα υδατά όμως καλύπτει και τις τρεις πτυχές. Αυτά ήταν τα διάφορα θέματα και τώρα θα δώσω το λόγο στον Στέφανη για τα ενδιαφέροντα ευρήματά μας. Ευχαριστώ πολύ Ρόπ. Περιέγραψες την εικόνα, ας περάσω εγώ στα ευρήματα. Πρώτα απ' όλα. Έχει μακρά ιστορία η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα τελευταία 40 χρόνια πολλά νομοθετήματα έχουν εισαχθεί εκτεταμένο πλέγμα ε, νομοθετημάτων έχει σαχθεί με διάφορες πτυχές. Ιδιαίτερα κορυφώνεται αυτή η προσπάθεια με την οδηγία πλαίσιο, με υψηλά επίπεδα ε, προδιαγραφών υγείας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, συλλογικό προγραμματισμό λογοδοσία, ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις για την ευέτευξη των στόχων και ούτω καθεξής. Πρόοδος. Ορατή και γρήγορη στην αρχή, με μείωση των επιπέδων ε, ρήπανσης στη δεκαετία του 80 και του 90 κυρίως. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε να περιορίζεται, να κάμπτεται η πρόοδος, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων υλοποίηση ε, τη οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι στόχοι τη οδηγία αυτή άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα υδάτινα οικοσυστήματα, το, το, τον, καθιστά τον τρόπο αυτό πιο περίπλοκο, τα βλέπουμε τα οικοσυστήματα με πιο περίπλοκο τρόπο και έτσι διαπιστώνουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι είχαμε κάνει αρκετά, ότι πρέπει να, να γίνουν πολλά ακόμα. Ε, άρα έχουμε ένα ποσοστό μόνο 80% που φτάνει στο επίπεδο το ικανοποιητικό προς το περιβάλλον, την επάρκεια, την καθαρότητα κτλ. Και όσο παρακολουθούμε την παρουσία χημικών στο ιδιάτινο περιβάλλον, κοκτέιλ χημικών, που είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί ως προς τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει και τις, ε, τον του στο οικοσύστημα. Επίσης έχουμε σημειώσει προβλήματα σε σχέση με τις ροές, την ταχύτερη ροή και την αστάθεια της ροής. Τα αποθέματα επίσης ε, δεν επαρκούν για να εξασφαλιστούν λειτουργούντα υγιή δηλαδή υδάτινα ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα. Μέτρα έχουν ληφθεί, αλλά δεν είναι αρκετά συνεπή, δεν φέρνουν το αναμενόμενο αποτελέσμα σχέση με, το, με τη δαπάνη και είμαστε σε μια κατάσταση ότι μπορούμε να περιγράψουμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός από φορέα. Μπορούμε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε ότι το προσχέδιο της Επιτροπής του λεγόμενου Blueprint προέβαινε σε μια εύρωστη και γενική αξιολόγηση και δεν σημειώνονται προβλήματα προς την αξιολόγηση αυτής της Επιτροπής. Τα στοιχεία που περιέγραψε ποιότητα, ποσότητα υδάτων και πτυχή χωρική πολιτικός σχεδιασμός και υλοποίηση, πώς, πώς σχετίζονται αυτά. Ξεκινώ λοιπόν με την ποιότητα. Στη θεωρία υπάρχει επιτυχής προσέγγιση, συνδυασμένη δηλαδή προσέγγιση με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας για το περιβάλλον και τις εκπομπές σε ευρωπαϊκό ή και εθνικό επίπεδο. Ανισορροπία όμως υπάρχει ως προς την χρήση των μέσων αυτών 50 διαφορετικά πρότυπα περιβαλλοντικά έχουν ε, εγκριθεί από τη θέση εφαρμογή, χωρίς όμως να ξεκινήσουν νέοι έλεγχοι εκπομπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο χάρη στην οδηγία. Και αυτό έχει να κάνει και με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, τα ζωτούχα, ε, που δεν αρκούν για να μειώσουν ε, την ρήπανση σε υδατινά Επίσης ε, η αναδυόμενη ρήπη, φαρμακευτικά κατάλοιπα και άλλη ρήπη όπως μικροπλαστικό και μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο φάσμα διαταρακτών. Το blueprint της Επιτροπής, το, προσχέδιο, το, το, το σχέδιο μελέτης, αναφέρεται σε κενά εφαρμογής και την επανεξισορρόπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των προδιαγραφών και των ελέγχων, στην ποιότητα των υδάτων νέα πρόκληση για όλες τις κοίτες ποταμών και όχι μόνο για τις ε, ε, λιγότερο έφορες περιοχές, τιμολόγηση και άλλα στοιχεία που όμως ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως και δεν έχουν καταστεί επαρκώς ε, χρήσιμα, άρα πολλά μένουν να γίνουν ως προς την ε, υλοποίηση σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης και πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα για το δεξιμό της κατανάλωσης. Εντοπίζουμε λοιπόν ευκαιρίες για καλύτερη ενσωμάτωση πολιτικής και σύνδεσμο ε, με την πολιτική για την αποτελεσματική χρήση των πόρων και πιο συγκεκριμένους στόχους και εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον προσδορισμό των στόχων. Το blueprint εστιάζεται στην ποιότητα όπως και στην ποσότητα ε, των υδάτων με κατευθύνες γραμμές ε, των οποίων όμως δεν βλέπουμε να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα. Πολλές από αυτές εξαρτώνται από την υλοποίηση της οδηγίας, παραμένουν όμως σε θελοντικό επίπεδο, παραμένουν θελοντικές και δεν βλέπουμε την επιβεβαίωση της χρήσης τους και την ε, εξασφάλιση αποτελεσμάτων ως προς το χώρο. Χωρική προσέγγιση και στοιχεία των υδάτινων οικοσυστημάτων από την οδηγία πλαίσιο. Έχουμε μόνο γενικούς δεσμευτικούς κανόνες και τη χρήση των ε, μέσων των τιμολογίων με την έννοια ότι φράγματα και το ε, χρησιμοποιη... Ε, καλύπτοντας προς το κόστος από εκείνους που τα χρησιμοποιούν. Στοιχεία όμως δεν υπάρχουν πάντοτε. Εμείς εντοπίζουμε δυνατότητες για περισσότερη ε, ολοκλήρωση της πολιτικής, πιο, αξιο... πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων και κυρίως κινητοποίηση χρηματοδότησης που είδαμε σε σχέση με τις ε, παιδιάδες όπου χρειάζεται παρέμβαση στο blueprint. Βλέπουμε να υπογραμμίζει ιδιαίτερος ε, το σύνδεσμο με την οδηγία τη σχετική με τις ε, πλημμύρες, με το πρασίσμα της ε, γεωργικής πολιτικής, και σε αυτό είναι σύμφωνο με, τις, με τη στόχευσή του. Στα ευρήματα λοιπόν, η υλοποίηση βλέπουμε να είναι αργή και ατελής η σχέση κοστος αποτελέσματος των μέτρων που εισάγουν τα κράτη-μέλη δεν είναι πάντα σαφής και θετική και βλέπουμε ότι είναι δύσκολο στη βάση αυτή να προσελκύεται χρηματοδότηση σε μεγάλη κλίμακα για τα μεγάλα έργα υποδομών που χρειάζονται. Διασύνδεση μεταξύ ε, σχεδίων διαχείρισης των ποταμών υπάρχει, κυρίως με τη λιωρική παραγωγή και τη διαχείριση πλημμύρα. Ε, υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ενσωμάτωση της νομοθεσίας για τις ρηπογόνες εκπομπές και βέβαια και τη πολιτική γενικότερα. προοπτικές στο μέλλον. Κοιτάζοντας προς τα προς, ορίζουμε τα κεφάλαια, τα θέματα, τη χρήση, τον οικοσχεδιασμό και τις μετρήσεις, τα φαρμακευτικά κατάλοιπα, για να αξιολογήσουμε το μίσο που θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αποδοτικότητα σε όρους κόστος αποτελέσματος. Δηλαδή περιορισμό της χρήσης των υδάτων και της ενέργειας με προδιαγραφές οικοσχεδιαστικές κυρίως για τις μπαταρίες βρύσης και το, τις κεφαλές ντους και την ε, ε, αλλαγή του διαθέσιμου ύδατος στα υδάτινα οικοσυστήματα πολιτικές και προγράμματα μέτρων ευρωπαϊκός συντονισμός για την αποκατάσταση των παιδιάδων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων υδάτινων στόχων, καλύτερα μέτρα για τον εντοπισμό φραγμάτων και υδατοφρακτών που ε, είναι πεπαλαιωμένα και που έχουν ξεπεράσει πια τον χρόνο ζωής τους και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα η ανανέωση αυτού του υλικού από κατάσταση κοιτών σε πολλά μέτρα βλέπουμε αποτυχία σε διαφορετικά στάδια γιατί υπήρξε αντίσταση από τον πληθυσμό και διάφορες ομάδες συμφερόντων πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση, διακυβέρνηση για να αποφεύγονται αυτές οι αποτυχίες συμμετοχή στα διαστρωτικά ταμεία, των διαστρωτικών ταμείων και ταμείων συνοχής για καλύτερη αποδοτικότητα, ενίσχυση των ε, εκπομπών ρήπων και μικρορυπογόνων ουσιών όπως φαρμακευτικών καταλήπων πρέπει να εξασφαλιστεί για την αποκατάσταση της ισορροπίας του του οικοσύστημα και την ε, ικανοποίηση των συνθηκών λειτουργία της οδηγίας πλαισίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο βεβαίως, ε, το οποίο όμως δεν έχουμε αναπτύξει διεξοδικά στην έκθεσή μας, ε, θα πρέπει να γίνονται αυτά. Βέβαια το εθνικό επίπεδο θα πρέπει να μελετηθεί χωριστά ασφαλώς. Τι προκύπτει από αυτά τα μέτρα που έχουμε περιγράψει. Σημειώνω και υπογραμμίζω ότι η δουλειά μας στηρίζεται σε εφιστάμενα στοιχεία και μόνο περιγράφει διάσταση. Δεν αποτελεί δηλαδή μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου της νομοθεσίας. Πολλές φορές είναι δύσκολο ή και ε, μη σκόπιμο να γίνει αυτή η μελέτη. Αλλά πολλά από τα αλλά πάνω απ' όλα πολλά από τα δεδομένα δεν είναι διαθεσή μας. καλύτερος τρόπος να μειώσουμε το κόστος και να ενισχύσουμε το όφελο είναι να υπάρχουν ελάχιστε προδιαγραφέ για την αποτελεσματικότητα κεφαλών του και ε, μπαταριών βρύση. Ε, μπορούμε χάρη σε αυτό, να αλλάξουμε τον οικοσχεδιασμό, δηλαδή να κερδίσουμε 2,6 δις το χρόνο για τα νοικοκυριά με αιτήσιο κόστος για την επένδυση σε 1,2 δισεκατομμύρια που πάλι θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά. Καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό χρειάζεται επίση για την αποκατάσταση των έργων ε, της παιδιάδας διάχυσης των ποταμών. Με υπολογισμό ε, ότι υπάρχουν 8,8 δις εκτάρια διαθέσιμα και βέβαια με τα στοιχεία που έχουμε από υφιστάμενες παιδιάδες της και τη δυνατότητα καλύτερης διατήρησης των υδάτων σε αυτές ώστε να περιορίζονται οι λοιπές ζημιές από τα ύδατα, καλύτερη παροχή ύδατος διάφορες άλλες χρήσεις ε, όπως ε, σε τουρισμό, αθλητικές εκδηλώσεις κτλ. Αυτό θα σήμαινε 39 δισεκατομμύρια εξοικονόμηση το χρόνο μέχρι το 2030. Εφόσον υπάρξει επένδυση με υψηλό κόστος ε, μέχρι το 2030, μέχρι το 2030 στα 362 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως για τις απαλωτριώσεις γης και τις ε, υποδομές που θα χρειαστούν. Όπως τα φράγματα υπερχείλησης. Περιορισμός της χρήσης ε, ύδατος και ενέργειας, ε, μεγαλύτερη δηλαδή αποτελεσματικότητα στην κατανάλωση ύδατος των οικοκυριών αφενός. Αυτό όμως θα πρέπει να έχουμε και υπόψη ότι η περιορισμένη κατανάλωση σημαίνει βράχη πρόθεσμα και υψηλότερες τιμές. Γιατί η φυστάμενη υποδομή δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Και έχει μια συγκεκριμένη ε, αναλογία κόστους αναμονάδα. Άρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ε, την διαφορά αυτή σε σχέση με τις ε, υφιστάμενες υποδομές και το κόστος. Δεδομένου ότι είναι παλαιά η υποδομή, είναι ενδιαφέρον να κάνουμε τη σχετική μελέτη. Η αποκατάσταση κοιτών υπερχείλησης ή παιδιάδων υπερχείλησης, βλέπετε εδώ για τον Δούναβη, μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει αρκετές χώρες και όπου προσπαθούμε να δούμε στο Δούναβη και τους παραποτάμους του 1,8 δισεκτάρια για την αποκατάσταση των σχετικών περίοδων υπερχείλησης με τη Γαλλία και, την, το Βέλγιο μαζί φτάνουμε στα 8,8 εκατομμύρια 2% των ε, υφιστάμενων γεών. Τελευταία μελέτη, ενίσχυση των ελέγχων εκπομπών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για μικρορύπαντες, μικρορύπους, ιδιαίτερα ε, φαρμακευτικά κατάλοιπα, με μέτρα που θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο εάν μπορούσαμε χάρη στον περιορισμό αυτών των καταλήπων στο ε, πλέγμα των υδάτων, στον υδάτων ορίζοντα, να περιορίσουμε τις συνέπειες. Βεβαίως, πρέπει να δούμε τι είδους ε, συστήματα μπορούν να εισαχθούν και τι είδους ε, διαφορετικά φάρμακα θα μπορούσε να σχεδιάσει η φαρμακοβιομηχανία το κόστος φυσικά του νέου αυτού σχεδιασμού να επηρεάζουν λιγότερο το ίδιο περιβάλλον. Για να καταλήξω, επιβεβαιώνουμε τις προκλήσεις που είχε εντοπίσει το blueprint της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε όμως μια διαφορετική εικόνα ως προς τις διαθέσιμες λύσεις. Υπάρχει δυνατότητα δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερη για τον περιορισμό των ρήπων. Υπάρχει δυνατότητα για περιορισμό της κατανάλωσης με ελάχιστες προδιαγραφές ως προς, ως προς την εσωτερική αγορά και η δυνατότητα για την αποκατάσταση των παιδιάδων υπερχείρησης ταμών. Αυτό νομίζω βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την αξιοποίηση των πόρων για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι μας. Σας ε, παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή μόνο τα κύρια ευρήματα. Πολλά είναι και τα παραρτήματα της μελέτης μας που ε, παρουσιάζουν ε, δεδομένα για τις διάφορες πολιτικές και το επίπεδο εφαρμογής τους και σας καλούμε να τα μελετήσετε. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now we can start uh, giving Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής μας. Ματίας Γκρότε πρώτος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Εγώ είμαι μεγάλος υποστηρικτής της οδηγίας πλαίσιο για τα έδατα που ξεκίνησε από το 2000 ε, και νομίζω ότι ο στόχος που και το 2000 ε, δεν έχει επιτευχθεί επαρκώς, απέχουμε πολύ αλλά πάλι και η υλοποίηση ε, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε πέντε κρατών μελών. Ε, είμαι ευγνώμων λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπω να επιμένει όχι για μια τυφλή εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και για παρακολούθηση και για συνδιαμόρφωση διαφορών διαδικασιών υλοποίησης. Και ξέρουμε ότι έχει μπορέσει, χάρη και σε διαδικασίες σε παραβάση, να επιτύχει ταχύτατη προσαρμογή των δημοτικών αρχών, οι οποίες μάλιστα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου χρειάστηκε να συνεδριάσουν με την προστασία των αστυνομικών αρχών προκειμένου να προστατευθούν από διάφορους ε, ε, αγριεμένους γεωργούς και άλλους που πίεζαν για κάτι το οποίο τελικά αφορούσε τα ευρωπαϊκά ύδατα. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγάλο πεδίο λοιπόν που αφορά και το Natura 2000 και πολλούς άλλους ε, ε, νόμους και νομοθεσία προστασίας. Και πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με δήμους που δεν έχουν στη θέση τους μέτρα, μέσα ούτε για την ε, αποκατάσταση ενός τετραγωνικού μέτρου εδάφους με βάση τους όρους αυτούς. Με βάση αυτά τα οποία ορίζει το Natura 2000 και η οδηγία πλαίσιο έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Θέλω λοιπόν ρητά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευαισθησία με την, και την, ε, για την ευαισθησία με την οποία και την ευφυΐα με την οποία διαχειρίστηκε το θέμα αυτό, γιατί είχε και τη βιομηχανία από τη μία να αντιμετωπίσει και τους γεωργούς. Και παρόλα αυτά κατάφερε να εξασφαλίσει πρόοδο σε μια κατάσταση δύσκολη. Όλα αυτά λοιπόν είναι αρκετά ενδιαφέροντα και συναρπαστικά. Και όπως είπα, δεν είναι πολύ φυσιολογικό να πρέπει να ζητήσουν ε, την προστασία της αστυνομίας οι δημοτικοί σύμβουλοι προκειμένου να εφαρμόσουν ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν έπρεπε ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, δύο συντάκτες της έκθεσης αυτής και πρέπει να πω προς τον συνάδελφό μου Ματίας ότι όπου έχουμε καλή νομοθεσία θα πρέπει να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας λέει επίσης πώς θα κάνει την νομοθεσία αυτή αποτελεσματική. εκτό τα σχόλια του κύριου Γκρότε. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε απάντηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η κυρία γιατί αυτή είναι τελικά η υπεύθυνοι για την εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας. Αυτή είναι, δεν αρκεί να έχουμε την νομοθεσία, πρέπει να επιβάλλεται αυτή η νομοθεσία, πρέπει να υλοποιείται η νομοθεσία. Ναι, προφανώ πρέπει να υλοποιείται από τα κράτη-μέλη, αλλά πολύ συχνά δεν υλοποιείται από τα κράτη-μέλη και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Και στην έκθεση αυτό ακριβώ βλέπουμε. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η τρίτη μου θητεία, είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε συνεχώ. Και πολύ συχνά λέμε ότι για παράδειγμα όσον αφορά τα ύδατα θα πρέπει να ξεφροτοθούμε μέσα 25 χρόνια όλες τις επικίνδυνες ουσίες. Ήδη από το 2015 έχουμε μία απόφαση στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία είναι κάπως πιο μετριοπαθής από αυτό το οποίο θέλαμε. Λέγεται απλώς να έχουμε μια καλή οικολογική κατάσταση όσον αφορά τα ύδατα. Ο αρμόδιος επίτροπος αλλά και η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπαν ότι η νομοθεσία αυτή δεν υλοποιείται στην πράξη, δεν έχει επιβληθεί στο σύνολό της από τα κράτη-μέλη. Έχουμε πολλά προβλήματα σε διάφορες χώρες όσον αφορά τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα ύδατα και βλέπετε ότι και οι υπουργοί περιβάλλοντος σε διάφορες χώρες πλέον φαίνεται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα επειδή πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένε νομοθεσίε για την υδατοκαλλιέργεια, για παράδειγμα. Και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί μια εντελώ παθητική στάση, τότε η μη εφαρμογή των ε, ευρωπαϊκών νομοθεσιών πολύ απλά θα συνεχίζεται. Δίνονται πολύ θετικέ συστάσει από τη μελέτη αυτή. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει τι προτίθεται να κάνει. Η μελέτη καλύπτει όλες τις πτυχές του ζητήματος. Θα ήταν πολύ καλό να ακούσουμε και κάποιες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μας έχετε δώσει επαρκείς απαντήσεις όσον αφορά την υλοποίηση της κοινωτικής νομοθεσίας. Ξέρω ότι ε, προβάλλει πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο τη μία πλευρά των πραγμάτων, το ότι δηλαδή νομοθετούμε, το ότι ε, δρομολογείται μια κοινοτική νομοθεσία, στην πράξη όμως θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία. Η μελέτη αυτή μας δίνει συγκεκριμένα συμπεράσματα και συγκεκριμένες συστάσεις. Θα ήθελα λοιπόν επακριβώς να μου πείτε κι εσείς, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να θεραπεύσετε την κατάσταση. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 το σύνολο της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως. Αν δεν κάνω λάθος λοιπόν έχουμε μπροστά μας κάποιες εβδομάδες μόνο. Εγώ θα σας έδινε ένα ολόκληρο χρόνο ακόμα. Αρκεί όμως να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα καταφέρετε να ελοποιήσετε αυτή την νομοθεσία. Νομίζω ότι οι απαντήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ικανοποιήσουν και τον κύριο Γκρότε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μιούλερ, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να εκφράσω τι ευχαριστίε μου για την παρουσίαση τη έκθεση που έλαβα μια κάποια καθυστέρηση και θα πρέπει επιμένω να τη μελετήσω προσεκτικά στι λεπτομέρειε τη. Δεν σα κρύβω ωστόσο ότι ω γεωργό στη Γερμανία έχω ήδη αντιμετωπίσει στα επιμέρου σημεία προβλήματα σχέση με την οδηγία πλαίσιο και τη γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, διαφορετικοί βαθμοί υλοποίησης και ελέγχου της υλοποίησης στα κράτη-μέλη. Για μένα λοιπόν Βεβαίω τίθεται το ερώτημα τι κάνει, την πράτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη μελέτη αυτή, τι θα ακολουθήσει και πώς όλοι αυτοί η διαθέσιμη οι, οι πόροι μπορεί να διατεθούν Και επίσης μιλήσατε για φράγματα υπερχείλησης στον χώρο του Δούναβη. Εγώ ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση εκεί με τα πόλτερς του Δούναβη, άλλωστε ζω στην περιοχή αυτή. Προτείνεται λοιπόν να συνεργαστούν οι αρχές με τους γεωργούς. Πώς μπορεί αυτή η γη να περάσει στην ιδιοκτησία των κρατών. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και βέβαια πάνω απ' όλα το θέμα της χρηματοδότησης. Ξέρουμε επίσης ότι είναι πολύ διαφορετικό ο τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιολογηθούν ε, τα σημεία μέτρησης στα διαφορετικά κράτη-μέλη, στα 28 διαφορετικά κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικοί ε, σταθμοί και κριτήρια Υπάρχουν λοιπόν κοινέ προδιαγραφέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε συμπαριλάβει κάτι τέτοιο στη μελέτη σας. Ή κοιτάτε μόνο τα δεδομένα όπως σας τα παρουσιάσαν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, and, uh, Σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο εσείς. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την ε, υπηρεσία ε, μας. Έχουν δουλέψει από ό,τι φαίνεται πολύ για το συγκεκριμένο πόνημα. Ένα ζήτημα μόνο με ανησυχίες ό,τι αφορά συγκεκριμένα την υποχρεωτική χρήση μετρητών νερού και κατά πόσον είναι και ουδέτερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας πλέον από τα κράτη-μέλη. Στη χώρα μου Έχουμε ένα πολύ προοδευτικό τρόπο χρέωσης ε, το τιμολόγησης του νερού. Ε, αυτό που λείπει νομίζω από την έκθεση είναι ε, το να έχουμε προσιτές τιμές ε, στο νερό. Θέλετε να έχουμε εξοικονομήσεις για τα νοικοκυριά, αλλά ζητάτε και ψηλότερες τιμές για να μην χρησιμοποιούν καταναλώνουν τόσο πολύ νερό οι συμπολίτε μας. Καλό είναι να αλλάξουν συνήθειες, αλλά με την εκπαίδευση οι πολίτες και όχι ε, να, να, το πετύχουμε τιμωρώντας τους, αυξάνοντας δηλαδή την τιμή του νερού. Γι' αυτό και καλωσορίζω και τις ε, ε για τη χρήση οικολογικών ε, συσκευών, μπαταριών βρύσης και τηλεφώνων ντους. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το πώς θα, βοηθήσει, ε, θα βοηθήσουμε την πολιτική, με την πολιτική για την ανάκτηση του κόστους να αλλάξουν το ε, Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, ε, στον Πάβελ Μίσικ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μας δώσει την άποψη της Κομισιόν σε σχέση με τη μελέτη αυτή. Good evening to everybody and thank you for the floor, Mr. Chairman. Uh, σας ευχαριστώ. Είμαι επικεφαλής της ε, ομάδας Αγία τα Ταΐδατα στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη κατά την άποψή μου και ιδίω η εκ των υστέρων αξιολόγηση που ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά ε, την ε, μέχρι τώρα κατάσταση εφαρμογή της οδηγίας. Ε, υποβάλαμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το Μάρτιο την έκθεση υλοποίηση, την έκθεση πεπραγμένου που αναλύουμε διάφορα σχετικά ζητήματα για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη που τους παρέχουμε συστάσεις και τα λοιπά και είναι παρόμοια τα ευρήματα με αυτά της έκθεση που μόλις παρουσιάστηκε. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκ των προτέρων ε, εκτίμηση για την ε, ανάγκη υλοποίησης κάποιων μέτρων, χαίρομαι που η μελέτη εστιάζει στους τομείς ε, για τους οποίους ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται η Κομισιόν και προτείνει πρωτοβουλίες, παραδείγματος χάρη χρήση του νερού, στρατηγική προσέγγιση για, τις, για τα φάρμακα, την ε, απορρίψη του στο περιβάλλον, για την πολιτική προϊόντων, ε, οικολογικό σχεδιασμό, επισήμανση. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη και η συγκεκριμένη έκθεση και τα στοιχεία της και τα συμπεράσματά της ε, θα μας δώσουν πολύτιμα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην μελέτη αντικτύπου των ελόγων πρωτοβουλίων. Σε ό,τι αφορά δύο άλλους τομείς, τη τιμολόγηση, μηχανισμούς τιμολόγησης, χρέωσης και τις ε, λεγόμενες ε, παιδιάδες ε, κατάκληση, την πλημμυρική κατάκληση. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνεται στη οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία για τις πλημμύρες. Εμέσως δε απαιτείται από τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους αυτές τις προσεγγίσεις στις δράσεις υλοποίησης. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έρχεται ε, σε μια πάρα πολύ σημαντική χρονική στιγμή αυτή η έκθεση. Είναι πολύ επίκαιρη διότι λύγει ο πρώτος κύκλος εφαρμογής Ξέρουμε ότι είναι εξαετή η κυκλοποίηση της οδηγία πλαίσια για τα έδατα. Είμαστε στο τέλο τη πρώτης περίοδου και στι αρχέ τη δεύτερη περίοδου και ακριβώ αυτή τη χρονική στιγμή τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν ε, τα δεύτερα σχέδια ε, διαχείριση των λεκανών απορροής. Ε, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί μέχρι τα τέλη του έτου οι στάσει και η έκθεση αυτή πιστεύω ότι μπορεί να τροφοδοτήσει τη διαδικασία αυτή αλλά και άλλε εκθέσει, άλλε δραστηριότητε εκτιμήσεις, μελέτες που θα πρέπει, ε, πιστεύω, ε, να βοηθήσουν και τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα εντοπίσουν. Θεωρούμε επίσης ότι η έκθεση αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί και στη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα που προβλέπεται για το 2019, αλλά ήδη έχουμε ξεκινήσει στα πρώτα βήματα, με πρώτο βήμα την αξιολόγηση των δεύτερων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής από την Κομισιόν που θα γίνει το 2016 και θα επακολουθήσουν άλλε ε, αξιολογήσεις, άλλε εκτιμήσει σχετικών πολιτικών. Θα δούμε πώς συμβάλλουν ε, στην εφαρμογή τη περιφερειακής πολιτικής, της ε, γεωργικής πολιτικής και επίσης θα ξεκινήσει και μια άλλη οικονομική αναλυτική μελέτη για την οικονομική αξία του νερού και των ε, υπηρεσιών ε, ίδρυυσης ε, για την οικονομία, ποιες είναι, ποια είναι τα ωφέλη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ύδατα και τι κόστος θα είχε η μία εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. Επομένως, τα απορίσματα της μελέτης σίγουρα θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, αν θεωρήσετε ότι αυτό θα ήταν σκόπιμο, θα μπορούσαμε να σας δώσουμε feedback εγγράφος, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια μεθοδολογικά ζητήματα και σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ε, κάποιων δεδομένων της Κομισιόν, αλλά αυτά είναι ίσον σημασία. Καταρχήν πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και επίσης οι συστάσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Και αφού μιλάμε για συστάσεις νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ αφενός των συστάσεων που απευθύνονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που μπορούν να εφαρμοστούν δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των εθνικών ε, αφετέρου συστάσεων. Γιατί αυτό που βλέπω εδώ ε, είναι ότι οι περισσότερες συστάσεις ε, προορίζονται για τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να υλοποιήσουν την υφιστάμενη και άκρος ικανοποιητική νομοθεσία για τα ύδατα. Καλό λοιπόν να φέρονται αυτά τα προβλήματα και υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη που προσπαθεί να ακολουθήσει μια πολιτική ισορροπημένη μεταξύ καρότη και μαστιγίου. Υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες επί παραβάση που είναι σε εξέλιξη ε, για κάποια κράτη-μέλη που παραβιάζουν τη νομοθεσία την Ευρωπαϊκή για τα ύδατα, αλλά υπάρχουν και κάποιες δραστηριότητες που στηρίζουν τα κράτη-μέλη στις προσπάθειες υλοποίησης των νομοθετημάτων αυτών. Αυτό που βλέπουμε, ίσως και πρώτη φορά, πιστεύω, είναι ότι γίνεται μια, ένας οικονομικός υπολογισμός ε, των επιπτώσεων της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας. Ε. Γιατί ένα από τα βασικά επιχείρηματα των κρατών μελών είναι ότι η υλοποίηση της οδηγίας αυτής ε, είναι δαπανηρή. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Αυτό το οποίο υπολογίζεται ως ετήσιο όφελο είναι πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και είναι υψηλότερο από το ποσό το οποίο επενδύουν ε, στη, ε, σε, τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή τη οδηγία για τα ύδατα και μάλιστα δύο και τρεις φορές σχεδόν. Αν χρησιμοποιήσουμε, αξιοποιήσουμε αυτή τη μελέτη και τι μελλοντικέ μελέτε που σχεδιάζουμε, θα μπορέσουμε πιστεύω να καταδείξουμε στα κράτη-μέλη ότι αποδίδουν οι επενδύσεις, ότι υπάρχουν οικονομικά και άλλα κοινωνικά ωφέλη από την επίτευξη των βασικών στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα για να είναι σε καλή κατάσταση τα ευρωπαϊκά ύδατα. Και αυτή η πολιτική δεν βελτιώνει απλά την ποιότητα ζωής, αλλά τονώνει στηρίζει και την οικονομία. Αλλιώς ε, συρρυκνούνται, περιορίζεται το οικονομικό και οικονομική ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν ε, ολοκληρώνω, αλλά αν θέλετε μπορώ να μιλήσω για μεμονωμένα μέτρα και συστάσεις. Αν θέλετε, παραλαμβάνω. Η Κομισιόν όμως, ε, ε αν θέλετε να σας πούμε τι μπορεί να γίνει για την υλοποίηση των συστάσεων της μελέτης. Μπορώ να σας πω κάποιες απόψεις, μπορώ να σας πω και κάποιες άλλες μας πρωτοβουλίες, όπως είναι η κοινή στρατηγική υλοποίηση, η στήριξη της καινοτομίας, πρόσβαση χρηματοδότησης για τα κράτη-μέλη και άλλου ε, φορείς και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you σας ευχαριστούμε. Οι συντάκτες ενδεχομένως της μελέτης πώ θέλουν να πάρουν το λόγο να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις ή να συνοψίσουν λίγο την συζήτηση ή θα μπορούσαν να σχολιάσουν αυτά τα οποία είπαν οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστούμε πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, το ζήτημα της χρήσης της γης, η πίεση που ασκείται όσον αφορά τη χρήση της γης, η ανάγκη αγοράς γης προκειμένου να αποκατασταθεί η γη αυτή. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και πολλές φορές διερωτάμε και ο ίδιος ποιος ποιο είναι το κόστος αυτό, το κόστος αγοράς της γης, το οποίο τελικά τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ ψηλό και δεν ξέρω αν θα πρέπει να απαιτείται κάθε φορά η αγορά γης από τους αγρότες προκειμένου να αποκατασταθεί στη συνέχεια το έδαφος και να συνδεθεί καλύτερα με το ποτάμι που περνάει από την περιοχή εκείνη. Και θα πρέπει ουσιαστικά να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αγρότες είναι μέρος της λύσης, ότι θα μπορούσαν και οι ίδιοι να αλλάξουν τον τρόπο που καλλιεργούν τη συγκεκριμένη γη και στα πλαίσια της, των σχεδίων αποκατάστασης των περιοχών που πλήττονται από πλημμύρε, θα μπορούσαμε ακόμα και να αλλάξουμε λίγο τους τρόπους της τοπικής οικονομίας, τους τρόπους που εφαρμόζεται η τοπική οικονομία. Να υπάρξει μια διαφοροποίηση δηλαδή ακόμα και στον τρόπο καλλιέργειας των εδαφών αυτών. Και θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από μια συγκεκριμένη δράση, γεωργική για παράδειγμα, και να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα πολυπλεύρως τις περιοχές αυτές. Ξέρετε ότι ε, αν δούμε την ε, προστασία, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι θέλουμε να καταργήσουμε κάθε οικονομική δραστηριότητα. Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Θέλουμε απλώ σε ορισμένε περιπτώσει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται μια συγκεκριμένη περιοχή, συγκεκριμένη εδάφη. Δεν μπορούσαμε εδώ πέρα να αναλύσουμε την κατάσταση και των 28 κρατών μελών. Επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένε περιπτώσει όσον αφορά την αποκατάσταση των περιοχών που πλήττονται από πλημμύρε. Επικεντρωθήκαμε κυρίω στο Βέλγιο, στο Δέλτα συγκεκριμένων ποταμών και είδαμε εκεί πέρα ποια είναι η υποδομή που υπάρχει προκειμένου να προστατευτούν οι περιοχές από τις πλημμύρες και είδαμε συγκεκριμένα στο Βέλγιο ότι η φυστάμενη υποδομή και η συντήρησή της ήταν πάρα πολύ ακριβή και κατάφεραν να βρουν εναλλακτικού τρόπους για να προστατεύσουν την περιοχή. Σε συνεργασία τώρα και με τη Γαλλία και με την γαλλική νομοθεσία την αποκαλούμενη Γκανέλ θα δημιουργήσουμε καλύτερα συστήματα και καλύτερες υποδομές για την προστασία των περιοχών που πλήττονται από πλημμύρε και ξέρετε ότι όσον αφορά τον Δούναβη ήδη πολλές σημαντικές δράσεις έχουν αναλυφθεί από την WWF. Μία ακόμα παρατήρηση όσον αφορά τις συστάσεις μας και όσον αφορά το εύρος του. τελικά να απευθύνονται περισσότερο στα κράτη-μέλη ή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στο λεγόμενο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι αναφερόμαστε εδώ πέρα και περισσότερο σε ευρωπαϊκέ κοινοτικέ παρεμβάσει όσον αφορά την τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, όπω για παράδειγμα για τον οικολογικό σχεδιασμό. Προφανώ το μέσο αυτό είναι κοινοτικό. Και επίση ισχύει η κοινοτική διάσταση όσον αφορά την αδειοδότηση των προϊόντων, όσον αφορά την αξιολόγηση τη τοξικότητα των προϊόντων, την αξιολόγηση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντικτύπου που μπορεί να έχουν ορισμένε χημικέ ή φαρμακευτικέ ουσίε. Νομίζω ότι όλα αυτά διευθετούνται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά την χωροταξική ανάπτυξη, και αναφέρομαι κυρίω εδώ πέρα στι περιοχέ εκείνε που πλήττονται από πλημμύρε, προφανώ εδώ πέρα η αρμοδιότητα είναι περισσότερο εθνική. Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να βρούμε αν υπάρχουν καλύτερε λύσει για τη διαχείριση των λεκανών απορροή ε, συγκεκριμένων ποταμών αλλά και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει μέσω των εργαλείων χρηματοδότησης ε, που διαθέτει. Ο Ρόμπ θέλει να πει για αυτός κάποια πράγματα. Ναι, όσον αφορά τη μέτρηση της κατανάλωσης νερού. Εμείς βασιστήκαμε σε κάποια στοιχεία που καταδεικνύουν τελικά ότι μειώνεται η κατανάλωση αν η πληρωμή γίνεται με βάση τη μέτρηση της κατανάλωσης του ύδατος. Αυτό είναι το βασικό μας ε, έβριμα και σε αυτό ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε. Και επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, μάλλον αν μειώσουμε τις περιπτώσεις διαρροής του ύδατος, μειώνεται και το κόστος. Ουσιαστικά θα πρέπει να περάσουμε από ένα σύστημα που έχουμε μία ελεύθερη, ανεξέλεγκτη παροχή ύδατος σε ένα σύστημα που ναι μεν θα παρέχεται ελεύθερο, ελεύθερα το νερό, αλλά που θα είμαστε σε θέση να μετρήσουμε πραγματικά την κατανάλωση, να αποσυντικοποιήσουμε την κατανάλωση του νερού. Επιφανειακά είδαμε κάποια στοιχεία, δεν έχουμε εξετάσει εντελεχώς το ζήτημα αυτό. Θελήσαμε όμως να δούμε με ποιου τρόπους θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε νερό και να μειώσουμε την κατανάλωση του ύδατος. Πάντως σχετικές μελέτες έχουν γίνει σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται χρόνος, αλλά πολλά κράτη-μέλη έχουν δει θετικά αποτελέσματα. Αυτά έχουμε να σας πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Όκεν θέλει το λόγο. Πάλι απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακολούθηση τι κάνετε σε σχέση με, την, με τα κράτη-μέλη. Παρακολουθείτε πραγματικά αν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό θα έπρεπε να κάνουν και αυτό θα έπρεπε να κάνετε και εσεί. Ας είμαστε λίγο συγκεκριμένοι. Φύσταται αυτή τη στιγμή μια οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Πέρα από τι συστάσεις, πέρα από τα όσα λέτε για, την, για τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, νομίζω ότι αν εφαρμόζαμε τη στρατηγική μας εδώ για τα ύδατα, θα είχαμε καταφέρει να πετύχουμε πολύ πιο θετικά πράγματα. Συγκεκριμένε συστάσεις υπάρχουν επίσης και στην κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα. Υποτίθεται ότι αυτή από το Σεπτέμβριο έπρεπε να εφαρμόζεται πλήρως. Στην πράξη όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Και η απουσία τελικά εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία, η απουσία Ευρώπη από όλα αυτά τα ζητήματα ουσιαστικά κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Όσον αφορά το ζήτημα της ύπαρξης φαρμακευτικών καταλήπων στα ύδατα, νομίζω ότι υπάρχει νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμόσετε πλήρως ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις αυτές. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις αυτές παρακολούθησης των κρατών μελών, ξέρετε ότι έχουμε εδώ πέρα μια συγκεκριμένη στρατηγική Καταρχάς, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, προσπαθούμε από κοινού να καταλήξουμε σε κάποιες ε, κατευθύντηρες γραμμές. Για τις χώρες όμως εκείνες που ε, δεν εφαρμόζουν σωστά την νομοθεσία, ξέρετε ότι υπάρχει διαδικασία επί παραβάση όταν ε, συνειδητοποιούμε ότι τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν παρακολουθούν σωστά την εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας, τότε ξεκινάμε μαζί τους κάποιες ε, συναντήσεις τεχνικής φύσεως, προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε καταρχάς κάποια πράγματα και ούτω καθεξής. Θέλουμε τώρα να δούμε μαζί με τα κράτη-μέλη πώς μπορούμε στα πλαίσια των διαχειριστικών τους προγραμμάτων να παρακολουθήσουμε καλύτερα την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και αναλόγως με βάση τα πορίσματά μας είτε θα εγκρίνουμε τη στρατηγική που ακολουθούν τα κράτη-μέλη, είτε θα μπούμε σε ένα νέο γύρο διαδικασίας επί παραβάση. Αν δούμε δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσει της οδηγίας. Όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, όντως υπάρχουν συγκεκριμένε υποχρεώσεις. Ο ίδιος ο νομοθέτης έχει επιβάλει συγκεκριμένε υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη, αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια για την ακρίβεια. Και εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάναμε μία προπαρασκευαστική μελέτη. Ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση, έγιναν και κάποια εργαστήρια με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και τώρα οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιες, όπως η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, προσπαθούν να δούνε ποια πολιτική θα ακολουθήσουν. Εξολογούμε τις διάφορες συναλλακτικές πολιτικές που έχουμε μπροστά μας και εξακολουθεί πάντως να εφίσταται αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία αναφερθήκατε και ελπίζουμε ότι πολύ γρήγορα θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε την πρωτοβουλία αυτή στην πράξη, πιστεύω μέσα σε ένα χρόνο. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Υπάρχει ακόμα μία βεβαιότητα σε επιστημονικό επίπεδο δεν έχουμε ακόμα αριστοκοποιήσει όλες τις ε, μεθόδους αξιολόγησης ε, του περιβαλλοντικού αντικτύπου, δεν έχουμε αναπτύξει πλήρως όλες τις μεθόδους παρακολούθησης για ορισμένες χημικές ουσίες ή ομάδες χημικών ουσιών. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς να προχωρήσουμε επισήμω σε μία ανακοίνωση η ομαδες χημικων ουσιων δεν μπορουμε λοιπον αυτη τη στιγμη εμεις να προχωρησουμε επισημως σε μια ανακοινωση η οποια θα μπορούσε στην πράξη να γίνει κοινοτική νομοθεσία και να εφαρμοστεί. Σε εσωτερικό όμω επίπεδο, ερχόμενοι σε επαφή με τα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία αναλαμβάνουν δράση, οι οποία ενδεχομένω να μην είναι απαραίτητα πλήρω αποτελεσματική, αλλά αποτελεί μια κάποια πρόοδο τελικά. Πολλά κράτη-μέλη αναλαμβάνουν δράση, έχουν ξεκινήσει συνεργασίες με διάφορα νοσοκομεία, προσπαθούν να ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα που έχουν για τα φάρμακα, για παράδειγμα, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν αρχίσει ορισμένα κράτη-μέλη να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες επεξεργασίας των υδάτων, λύσεις οι οποίες βέβαια είναι πολύ ακριβές, αλλά έχουν επιλογή από ορισμένα κράτη-μέλη. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με τα κράτη-μέλη, συζητάμε μαζί τους και προσπαθούμε από κοινού να δούμε πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περισσότερο τις βέλτιστες αυτές πρακτικές και σε άλλα κράτη-μέλη. Πώς μπορούν δηλαδή να αποφεληθούν ορισμένα κράτη-μέλη από πολύ θετικές εμπειρίες που είχαμε στη Γερμανία, τις κάτω, τις κάτω χώρες στη τη Γερμανία. και στη συνέχεια θα μπορέσουμε εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναπτύξουμε ένα σύστημα αξιολόγησης αντικτύπου και να προχωρήσουμε σε μία επίσημη νομοθετική πρωτοβουλία. Μολονότι μπορεί να μην φαίνεται στην πράξη ότι έχει γίνει κάτι σημαντικό, στην ουσία έχουμε ξεκινήσει μια πολύ σημαντική προεργασία με τα κράτη-μέλη προκειμένου να διηγηθούμε μια μέρα σε μια κοινοτική ξεκινησει μια πολυ σημαντικη προεργασια με τα κρατη μελη προκειμενου να οδηγηθούμε μια μερα σε μια κοινοτικη πολιτικη και παράλληλα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν αυτά σε εθνικό επίπεδο, εθνική δράση. Και όπου συναντάνε προβλήματα προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Οπότε και ξανασυνεδριάζει η Επιτροπή Ένδυση 9 το πρωί. Γεια σας.